ψηφοφοριών πρώτα απ' όλα. Θέλω να σας αναφέρω ότι η προθεσμία για την κατάθεση <clears throat> τροπολογιών στο Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013 έχουν θεσπιστεί με συμφωνία της Επιτροπής Προϋπολογισμού ως εξή Για τις επιτροπές και τους, τις ομάδες ή τουλάχιστον 40 βουλευτές 6 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. 5η 6 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι για τις πολιτικές ομάδες 13 Δεκεμβρίου στις 12. Θέλω επίσης να κάνω μια δήλωση εξ του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, στην